Um, Καλώς ορίσατε όλοι ε, στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Χαίρομαι που βλέπω μερικούς βουλευτές παρόντες. Αρχίζουμε λοιπόν. Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε την Κροατική Προεδρία που θα μας μιλήσει σήμερα το απόγευμα. Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα την περασμένη εβδομάδα να έρθω στο Ζάγκρεπ, αλλά άκουσα από τον αντιπρόεδρό μας κύριο Λαγκοντίνσκι πόσο χρήσιμη και γόνιμη ήταν η συζήτηση. Είδατε στον τρίτο τριμερή διάλογο πόσο δραστήρια ήταν η Κροατική Προεδρία πριν από δύο εβδομάδες και προετοιμάζει και τον αυριανό τριμερή διάλογο. Και φυσικά ε, μας ενδιαφέρει να ακούσουμε περισσότερο για τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σας δίνω μέσω στο λόγο για την εισαγωγική σας παρουσίαση και μετά θα ακούσουμε και ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Νομικής Επιτροπής, με χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης. Είναι μια περίοδος η οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές δυσκολίες. Το σλόγγαν της Προεδρίας μας είναι μια ισχυρή Ευρώπη στην εποχή των προκλήσεων τέσσερις προτεραιότητες. Πρώτα, μία αναπτυσσόμενη Ευρώπη. Δεύτερον, μια Ευρώπη η οποία ενώνει, δεύτερον, τρίτον μάλλον μια Ευρώπη που προστατεύει και τέταρτον μια Ευρώπη φάρος στον κόσμο. Αυτές είναι οι προτεραιότητες λοιπόν για μας ιδιαίτερα στον κλάδο της προστασίας των πολιτών από την Ευρώπη. Θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας ε, για το μέλλον του χώρου ελευθεριών, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Στα πλαίσια μιας στρατηγικής συζήτησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια της συζήτησης για τα επιμέρους θέματα των εσωτερικών υποθέσεων και της δικαιοσύνης, προηγήθηκαν συζητήσεις και κατά τη διάρκεια της Ρωμανικής και κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε το επόμενο πενταετές θα έλεγα πρόγραμμά μας. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν προς συζήτηση και στην άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης ε, στο Ζάγκρεμπ στις 24 Ιανουαρίου η ανάγκη καθορισμού των στρατηγικών επιλογών για τον τομέα της ασφάλειας και των ελευθεριών είναι ευθύνη την οποία μας δίνει η ίδια η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ξεκίνησε από το 1989, μετά το 2004, το 2009 στη Στοκόλμη και το τελευταίο πρόγραμμα στρατηγικό για τις εσωτερικές υποθέσεις και τις ελευθερίες είναι του 2014. Το τελευταίο μάλλον πρόγραμμα υιοθετήθηκε τον προηγούμενο Ιανουάριο. Περιλαμβάνει συγκεκριμένα επιμέρους στοιχεία απαραίτητα για τον χώρο της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και των δικαιωμάτων. Η κροατική προεδρία δεν ξεκινά από μηδενική βάση, εκμεταλλεύεται τις ε, συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει για τα θέματα της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαριστούμε γι' αυτό τους υπόλοιπους της Τρόικα, δηλαδή Ρουμανία και Φιλανδία. Η βασική ιδέα είναι να μπορέσουμε να εργαστούμε στα διαμεθοριακά θέματα που είναι θέματα που αποτελούν πρόκληση για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Θα πρέπει να εμείνουμε στους τρόπους με τους οποίους θα επικοινωνούμε. Προβλέπουμε μία δομή για το μέλλον η οποία εδράζεται στις αξίες, τις βασικές αρχές της Ένωσης και την προστασία του κοινού ευρωπαϊκού χώρου και μέσω των νέων τεχνολογιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης της Ζαγκάμπρια, κάνουμε προτάσεις για τις νέες στρατηγικές οι οποίες θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν και τις δικές σας προτάσεις. Τον Απρίλιο, στα πλαίσια του Κορεπέρ, θα κάνουμε ε, μια συζήτηση για τις στρατηγικές αυτές ε, ε, γραμμές έτσι ώστε να συζητηθούν επίσημα από το Συμβούλιο και να πάρουμε το πράσινο φως του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τένος του μητός Μαρτίου. Να υπογραμμίσω ότι η κρατική προεδρία είναι σε μόνιμη επαφή με την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτό έτσι ώστε οι κατευθυντήριες γραμμές να υιοθετηθούν επί, τη βάση την οποία, επί της βάσεως την οποία προανέφερα. Για τα θεμελιώδη δικαιώματα η Κροατία θα ε, υπερασπιστεί την σημασία που έχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τους εσωτερικούς κανόνες. Ήδη από το 2018 επικύρωσε η χώρα μου τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, για τη βία εις βάρος των γυναικών και την οικιακή όπως λέγεται βία έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή διάκρισης και κάθε μορφή βίας εις βάρος των γυναικών. Η καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών είναι πάντα βασική προτεραιότητα της Προεδρίας μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σχετικά τώρα με τα οικονομικά προγράμματα, <clears throat> τα χρηματοδοτικά, συγγνώμη, εμείς θα κλείσουμε τη συζήτηση για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων δικαιοσύνη, δικαιώματα και αξίες, όπως είχαμε αποφασίσει και στα πλαίσια των προηγούμενων συναντήσεων. Γενικά, γύρω από το ποινικό, θα προωθήσουμε συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα και για τις διαδικτυακές αποδείξεις και θα φροντίσουμε έτσι ώστε ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας να αναλάβει τις ευθύνες του το ταχύτερο δυνατόν και θα κάνουμε μία συνάντηση στο σπλή τον μήνα Απρίλιο. Η Προεδρία θα συγκεντρώσει την προσοχή της στις προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού για τη γνωστοποίηση των πράξεων αναχώρα, όπως επίσης και για την πρόταση ψηφίσματος για την απόκτηση αποδείξεων πριν από το τέλος της δικής μας Προεδρίας. Θέλουμε να κάνουμε και βήματα πρόοδου σε άλλους τομείς, όπως η πρόταση η οποία έχει σαν στόχο ε, η, αμφ, η αμφισβήτηση των εκχωρήσεων χρεών. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα μπορέσουμε να συζητήσουμε στα πλαίσια των επαγγελματικών ε, δικτύων όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε επίπεδο αστικού δικαίου. Για να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η Κροατική Προεδρία θα προχωρήσει με το σύστημα e-justice χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη σχετικά για την ε, κατάρτιση και την εκπαίδευση των ε, στελεχών του δικαστικού σώματος. Έχουμε τέσσερις προτεραιότητες. Μία από τις προτεραιότητες αυτές τις επιμέρους είναι η κάλυψη του συνόλου του χώρου της δικαιοσύνης, ε, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε αυτό που ονομάζουμε μια προστάτηδα Ευρώπη, μια Ευρώπη που προστατεύει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί μόνο σαν χώρος ελεύθερης διακίνησης, αλλά σαν χώρος που σέβεται τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα βοηθήσουμε στην σωστή κατάρτιση των δικαστών, των δικαστικών συμβούλων, ανακριτών κτλ. έτσι ώστε να διευκολυνθούν ε, στην καθημερινότητά τους. Αυτό θα επηρεάσει άμεσα με τη σειρά του την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και θα βοηθήσει την προστασία των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Η κατάρτιση λοιπόν των μελών του δικαστικού είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει στην ημερήσια διάταξη και στις συζητήσεις με τους πολιτικούς υπευθύνου, από τα κράτη-μέλη αλλά και από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δικαστική συνεργασία είναι ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην ανεπίσημη συνάντηση του Συμβουλίου τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησαν τις απόψεις τις οποίες έχουν έτσι ώστε να αποδείξουν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μην εξαιρεθεί καμία κατηγορία εργαζομένων στον τομέα του δικαίου από τις ε, μορφές και τις δυνατότητες κατάρτισης. Έτσι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα αποκτήσουμε όλες τις απαραίτητες ε, ε, γνώσεις. Τώρα, ε, για τον προγραμματισμό των υπουργικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Όπως είπα στο παρελθόν, έγινε μια πρώτη ανεπίσημη συνάντηση στον τομέα της δικαιοσύνης στις 23 Ιανουαρίου στο Ζάγκρεμπ. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα οργανώσουμε δύο επίσημες συναντήσεις του Συμβουλίου, 12 και 13 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και α, ε, επίσης 5 ε, και 6 Ιουνίου. και στο τέλος του Μαΐου θα υπάρξει και η συνάντηση με τις Ηνωμένε Πολιτείες του Ντουμπρόβνεκ. Ευχαριστώ τα μέλη. Ε, Madame Sorry. Ε, κυρία Βόλαχ, έχω μια ερώτηση για τη διαδικασία της επιτροπολογίας πώς θα συνεχιστεί, χωράει στο εξάμεινό σας. Πώς το βλέπετε εσείς από πλευράς Προεδρίας. Να πω δύο λόγια για τη διαδικασία αυτή καθ' αυτή. Το 2017 πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρηση της επιτροπολογίας και η τελευταία συνεδρίαση, Γιούρι, ε, ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Επανέρχεται συνεχώς το ζήτημα ε, για το πώς πλαισιώνει τα νομοθετήματα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταλήγουμε πάντα στην Επιτροπολογία. Τα κράτη-μέλη δεν γνωμοδοτούν και είναι πολύ κρίμα αυτό, ιδιαίτερα ε, όταν πρόκειται για ευαίσθητους τομείς του δικαίου και καλό θα ήταν τα κράτη-μέλη να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες. Αντιθέτως, πολύ συχνά βλέπουμε να απέχουν τα κράτη-μέλη και ε, στη συνέχεια δηλώνουν ότι ψήφισαν διαφορετικά. Ε, αυτό δεν βοηθάει στην τόνωση της φήμης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των πολιτών. Θα πρέπει ο κανονισμός του 2011 επιγόντως να αναθεωρηθεί. Η ομάδα μας, σοσιαλιστές και δημοκράτες, αλλά ελπίζω και οι άλλοι συνάδελφοι να συμφωνούν. Θέλουμε να δοθεί συνέχεια και να δείξουμε ότι τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπλοκάρει, αλλά αυτός που μπλοκάρει είναι το Συμβούλιο και δεν μπορεί να συμφωνήσει και ε, ρωτώ την Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου. Ποια είναι η στρατηγική σας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας για να αποτελματωθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο τα πράγματα είναι σε ένα νεκρό σημείο. Έχετε προτάσεις για να εγκριθεί ε, έτσι μια γενική θέση στο Συμβούλιο. Δική μου ελπίδα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ακολουθήσει κάποιες φωνές που ακούμε εδώ στο Κοινοβούλιο και αποσύρει την πρότασή της. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο το οποίο απέφχομαι, τι θα γίνει, εσείς θα υποστηρίξετε νέα πρόταση. Φοβάμαι ότι θα είναι μια αποδυναμωμένη ε, εκδοχή της τρέχουσας πρότασης. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς το βλέπει η Προεδρία και τι θέση λαμβάνει σχετικά. Hvala lijepo na ovom Μια ερώτηση ήθελα να υποβάλω. Επίσης σχετικά με την επιτροπολογία. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις στις ομάδες εργασίας. Ε, θα εξακολουθήσουμε να δουλεύουμε ε, για το θέμα αυτό. Έχουν υπάρξει επίσης διαπραγματεύσεις ε, στα πλαίσια ε, του Συμβουλίου τον μήνα ε, Ιανουάριο. Η ΔΕ Προεδρία θα συνεχίσει να εργάζεται έτσι ώστε να προωθήσει το θέμα αυτό, τον φάκελο αυτό κατά τη διάρκεια της Κροατικής Προεδρίας. Σας διαβεβαιώ ότι η Κροατική Προεδρία θα συνεχίσει την εργασία στα πλαίσια των ομάδων εργασίας έτσι ώστε να επιτευχθεί η θέση. Ο κύριος Ράντεφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα καταρχά να σας ευχηθώ καλή τύχη. Ε, καλή τύχη στην Προεδρία σας για το επόμενο εξάμεινο. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες σας για τον τομέα της δικαιοσύνης. Λέτε ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες στη δικαστική ποινική συνεργασία θα είναι να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος και να εγκριθεί ο κανονισμός Ε, για την πρόσβαση σε έγγραφα, δικαστικά και εξοδικαστικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, για να συνοηθούμε και να συντονιστούμε στα κράτη-μέλη σε θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο για τη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία. Η αγαστή συνεργασία των δικαστηρίων είναι εκ των όνου κάνευ για να λειτουργεί σωστά εσωτερική αγορά. Το 2018 περίπου 3,4 εκατομμύρια αγωγές ε, κατατέθηκαν σε αστικό και εμπορικό δίκαιο ε, με διασυνοριακό χαρακτήρα και πολλές φορές χρειάζονται εκεί αποδεικτικά στοιχεία από ένα άλλο κράτος μέλος. Και ο σχετικός κανονισμός προβλέπει κάποια μέτρα ε, διευκόλυνσης πρόσβασης στα στοιχεία αυτά. Εγώ νομίζω ότι η προστασία των βασικών θεμελιδών δικαιωμάτων, προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει ε, ε, τη διασυνορική συνεργασία, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ελπίζω να είναι γόνιμη η συνεργασία μας. Εξ ονόματος του συντονιστού μας, του κυρίου Φως, έχω να θέσω ένα σημαντικό ζήτημα. Το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ψήφισμα με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νομική προστασία ενηλίκων. Υπάρχει μια σύμβαση της Χάγης σχετικά του 2000 για τη διεθνή προστασία ενηλίκων. E, Απάντηση. Όντως, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όσον αφορά την επίδοση των ε, πράξεων ε, πρέπει να προχωρήσουμε γιατί πρόκειται για θέματα και κείμενα πάρα πολύ σημαντικά. Ε, το κείμενο σχετικά με την επίδοση, τη σωστή επίδοση των εγγράφων διευκολύνει ε, την ε, σωστή πρόθεση των διαδικασεών, ε, την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των εμπλεκομένων και επομένως μέσω αυτών των στοιχείων μπορούμε να φτάσουμε σε απόδοση της δικαιοσύνης που θα γίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Εμείς θέλουμε επίσης να εξυγχρονίσουμε το θέμα της δικαστικής συνεργασίας και άλλωστε αυτό αποτελεί και έναν από τους ε, κύριους στόχους και τις προτεραιότητες της κρατικής Προεδρίας. Τον μήνα Δεκέμβριο του 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε ε, θέση. Βέβαια για την ώρα ε, συζητούν τη θέση αυτή ε, οι διάφορες ομάδες εργασίας. Επίσης υπάρχει το ζήτημα του παραρτήματος γιατί και σε αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε. Τα παραρτήματα είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά την υλοποίηση του κειμένου. Ε, σήμερα θέλουμε να επιτύχουμε πλέον και τεχνική εναρμόνιση των τροποποιημένων ε, κειμένων. Η Προεδρία είναι στην ευχάριστη θέση να σας πει ότι ο τριμερής διάλογος με το ε, Κοινοβούλιο θα ξαναρχίσει ως ο Ευχαριστούμε ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο ε, γιατί είναι διατεθειμένο να ξαναξεκινήσει τον ε, διάλογο όσον αφορά κυρίως το αστικό ε, δίκαιο. Πρόθεση της Κροατικής Προεδρίας είναι να κλείσει τους τριμερείς διαλόγους όσον αφορά τα δύο ζητήματα που αναφέραμε προηγουμένως και με τον τρόπο αυτό να προωθηθεί η επικαιροποίηση, εξυγχρονισμός και ψηφιοποίηση Τη της ε, δικαιοσύνης. Είναι πολλές όντως οι υποθέσεις ε, και επομένως οι επιλύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι καλή τύχη στις μελλοντικές σας ε, ε, αρμοδιότητες. Ε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και για την Ρουμανία. Πρώτα απ' όλα όμως να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά το πολυσυζητημένο θέμα της ε, κατάστασης δικαίου, του κράτους δικαίου, κυρίως ε, σε σχέση ε, και σε συνδυασμό με την πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους. Δηλαδή, εάν και εφόσον υπάρχει παραβίαση του κράτους δικαίου, θα πρέπει να σταματήσει και η ροή ευρωπαϊκών, των ευρωπαϊκών πόρων. Θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή αντίληψη για το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τούτη τη στιγμή είναι δύσκολο να ξεκαθαριστεί κανείς και να δώσει ένα ξεκάθαρο ορισμό αυτού του μηχανισμού. Και να σας κάνω και μια ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το ενδεχόμενο κύρωσης των πραγματικών... Ε, ε των πραγματικών δικαιούχων των πόρων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πρόκειται για δημόσιε ε, αρχέ, είτε για ιδιωτικέ ε, αρχέ, ε, αυτοί δεν μπορούν να κυρωθούν μέσα ω ως τελικοί δικαιούχοι και όλα αυτά βέβαια ε, με νόμιμο τρόπο. Από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε ευρωπαϊκά χρήματα σε χώρες στις οποίες υπάρχει ε, παραβίαση του κράτους δικαίου. Δεύτερον, θέλω να αναφερθώ ε, στην ένταξη της Ρουμανίας στην ζώνη Σέγγεν όλες οι αρχές λένε ξεκάθαρα ότι η Ρουμανία πλέον ε, έχει όλα τα κριτήρια, καλύπτει όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να ε, ε, ενταχθεί στον χώρο Σέγγεν. Ωστόσο και παρόλα αυτά το Συμβούλιο Ε, μέσω κάποιας σειράς κρατών μελών δεν ενδιαφέρονται να αποδώσουν δικαιοσύνη στους Ρουμάνους πολίτες που δεν μπορούν να ε, ε, έχουν αυτήν την πλήρη ελευθερία κυκλοφορίας αγαθών και ατόμων και προσώπων όπως ισχύει για τους άλλους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση όσον αφορά το κράτος δικαίου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω ε, αυτά τα οποία αναφέρονται στο στρατηγικό πρόγραμμα. Ε, υπάρχουν κοινέ αξίες όπως είναι η δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος ε, δικαίου που αποτελούν τα στοιχεία από των οποία εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση παραβίασης η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να λαμβάνει ε, δράση και μέτρα. Εμείς κατά τη διάρκεια της κρατικής προεδρίας αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία ε, στο σημείο αυτό και επομένως θα υπάρξουν στρατηγικές στρατηγικές γραμμές όσον αφορά τον χώρο δικαιοσύνης και ελευθερίας ε, εμείς θέλουμε να προωθήσουμε ε, τις ε, θεμελιώδεις αξίες αλλά και να προωθήσουμε και το διάλογο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοούμε βεβαίως ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά ορισμένες χώρες και θεωρούμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να μελετηθούν. Ε, θα ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά ε, μέσω του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ε, η κροτική Προεδρία. Και θα προβλεφθούν νέοι μηχανισμοί, μάλλον πριν εφευρεθούν νέοι μηχανισμοί κυρώσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους και στα όρια τους οι ισχύοντες περιορισμοί. dok Επίσης, όσο δεν ε, ε, υπάρχει συμφωνία σε υψηλό επίπεδο, η Κροατική Προεδρία θα συνεχίσει τις προσπάθειες. Εάν προκύψει συμφωνία ε, σε υψηλό επίπεδο και κυρίως στα πλαίσια του πιδελταπή θα χρησιμοποιηθεί ε, το κουτί των διαπραγματεύσεων ε, για να συνεχιστούν οι εργασίες, κυρίως όσον αφορά τον κανονισμό για το κράτος δικαίου. Πρέπει να πω ότι για το κράτος δικαίου υπάρχουν και κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ε, εκαλύφθησαν υπό Ρουμανική Προεδρία. Είναι όμως πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινή αντίληψη, συναντήληψη όσον αφορά ε, όλων των θεμάτων στα πλαίσια του προγράμματος ε, δικαιοσύνη, δικαιώματα, αξίες. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μηχανισμός συγκεκριμένος στόχος του οποίου θα είναι η προστασία των δικαιωμάτων και η ευαισθητοποίηση των πάντων όσον αφορά τα θέματα αυτά, ευνοώντας ακριβώς την καλή εργασία της κοινωνίας των πολιτών, των διασυνοριακών οργανώσεων, ε, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών κλπ. Έτσι ώστε να διασφαλιστεί το κράτος δικαίου. Ε, και ε, με τον τρόπο αυτό να ενισχύσουμε τη δημοκρατία αλλά και τη διαφάνεια εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Κύριος Λαγκοντίνσκι. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Ντράζεν, ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την Προεδρία σας. Είχαμε και εξαιρετική συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, όπου ε, είχα την ευκαιρία εκπροσωπώντας την Επιτροπή ε, Γιούρη να δω πόσο καλά ήταν οργανωμένη η συνάντηση αλλά και πόσο ουσιαστική ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Τρία ερωτήματα έχω να θέσω. Πρώτον, το συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα και οι Υπουργοί Δικαιοσύνη σε βάθος αυτό το θέμα όντω του κράτους δικαίου κατά τη διάρκεια αυτής τη συνεδρίασης. Τι έλειπε όμως, ε, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Υπουργών Δικαιοσύνη. Ήταν η θέση της Προεδρίας για τη διαδικασία του άρθρου 7. Όπω γνωρίζετε, ε, έχουμε δύο προσφυγές αυτή τη στιγμή βάση του άρθρου 7, πράγμα που ανησυχεί πολύ τους ευρωβουλευτές. Τι θα γίνει το επόμενο εξάμεινο. Συγκεκριμένα, και ακριβώς. Εσείς πώς βλέπετε το ρόλο σας στην προώθηση αυτής της διαδικασίας για το άρθρο 7 και πώς προτίθεστε να ε, συμπεριλάβετε το κοινοβούλιο που έχει εμπνευστεί όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης, ε, μεγάλο θέμα στη συζήτηση και στο πρόγραμμά σας ε, καλύπτει το θέμα της, της κατάρτισης των ε, δικαστικών λειτουργών. Μόνο για δικαστές ε, θα έχετε ε, εκπαίδευση για δικαιώματα ΛΟΑΔ, αντισημιτισμό, αντιτσιγκανισμό κτλ. Που θα πρέπει να εκπαιδεύονται και οι δικαστικοί και οι αστυνομικοί. Και το τρίτο είναι χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων για το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη αλλά και τη Eurojust. Όπως θυμάστε το συζητήσαμε γι' αυτό και ε, ανησυχούσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποχρηματοδότηση του Eurojust. Έχετε συγκεκριμένα σχέδια. Πρώτον, συμφωνείτε και δεύτερον, πώς προτίθεστε να βελτιώσετε την κατάσταση όπου υποχρηματοδοτείται η Eurojust σε σύγκριση με τη Europol ή τη φύλαξη των συνόρων, όπως έχει σχεδιαστεί για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ε, ε, φυσικά τα συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα και τα αναλύσαμε και τις δεξιότητες και ε, τα προσόντα των δικαστικών και τη διαδικασία βάση του άρθρου 7. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι θα πρέπει όλοι να εξαντληθούν πριν προχωρήσουμε σε κυρώσεις και θα πρέπει ε, να επενδύσουμε όλη την ενέργειά μας στο διάλογο για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα ουσιαστικό. Και από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα, θα δούμε την επόμενη φάση. Ε, τώρα, για το διάλογο στο ιστορικό του Συμβουλίου. Το Νοέμβριο αποφασίσαμε να ενισχύσουμε την προσέγγιση μας, δηλαδή ε, ε, να χρησιμοποιούμε διάφορες πηγές. Θα υπάρξει και μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου με ένα κατάλογο όλων των θετικών και αρνητικών τάσεων στα κράτη-μέλη ε, για την κατάρτιση και εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών και λοιπόν υπαλλήλων. Στο Ζάγκρεπ το συζητήσαμε, αλλά και την ανάγκη να εξυγχρονιστεί η δικαιοσύνη και να επιμένουμε περισσότερο στην επαγγελματική εξέλιξη και στα διοδρομία ε, των δικαστικών και όλα τα θεσμικά όργανα ε, φυσικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχουν θέση για όλα αυτά που αναφέρατε στο δεύτερο θέμα. Στο τρίτο τώρα, τη χρηματοδότηση. Στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχω να σας απαντήσω αυτό που απάντησα και στην προηγούμενη ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, οι αρμοδιότητες της Προεδρίας είναι αρκετά περιορισμένες θα πρέπει πρώτα να ληφθεί η απόφαση στο υψηλότατο πολιτικό επίπεδο, στο Συμβούλιο ε, Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μετά εμείς θα συζητήσουμε την εφαρμογή. Ευχαριστώ. <clears throat> <clears throat> Ε, ε, Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. sobre divulgación de información sobre Το θέμα είναι ακριβώς τι γίνεται με τις εκτίσιες εκθέσεις αναχώρα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η ανικανότητα για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα είναι κάτι το οποίο εντυπωσιάζει και είναι κάτι το οποίο ε, θέτει σε αμφισβήτηση αν οι ικανότητες των Βεξελών είναι τέτοιες για να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες της, για ε, των θεμάτων τα οποία έχουμε επιλέξει και να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε το μπλοκάρισμα της κατάστασης και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα νομικά άλοθη σύμφωνα με τα οποία η νομική βάση της συμφωνίας ε, δυστυχώς αυτά χρησιμοποιούνται για να αποκρύβουν την αποτυχία την ανικανότητά μας να ε, έχουμε να λειτουργήσουμε, ε, να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις και αυτό να το κάνουν φυσικά βασικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Θα ήθελα την επίσημη θέση της κυβέρνησής σας. Έχετε και εσείς την υποχρέωση θα έλεγα να ξεπεράσετε αυτό το μπλοκάρισμα και να δώσουμε στην κοινή γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια συμφωνία ικανοποιητική. θα πρέπει να σταματήσουν τα κράτη-μέλη να αποκρύβουν α, τις πραγματικές αιτίες για την α, μη διαφανή, αν θέλετε, αντιμετώπιση των α, πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Hvala lijepo na ovom pitanju. Moram reći da su ove pravne rasprave o pravnim... Αυτές οι συζητήσεις γίνονται για την νομική βάση, ε, όπως επίσης και για τις διαδικασίες γενικά έχουν μεγάλη σημασία. Η κρατική Προεδρία συνειδητοποιεί τη σημασία που έχουν τέτοια θέματα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικά για το κοινό. Για το κοινό. Το πρόβλημα όμως τίθεται πάντα για τη νομική βάση της πρότασης και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λύσουν τα κράτη-μέλη. Η Κροατική Προεδρία σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και σε συνεργασία με τις νομικές τους υπηρεσίες προσπαθούν να βρουν μία λύση. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου εκφράζει την άποψη ότι οι νομικές βάσεις θα πρέπει να βασίζονται στο 115 και όχι στο 50 όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε θα πρέπει στο Συμβούλιο να υπάρξει ομόφωνη απόφαση για την αλλαγή της νομικής βάσης. Μια τέτοια ομοφωνία δεν υπάρχει. Το θέμα των νομικών βάσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί διαφοροποιούνται τα πράγματα ανάμεσα στο άρθρο 50 και στο άρθρο 115 για το αν θέμα λογιστικών προτύπων ή αν θέμα φορολογικό κυρίως. Απαιτείται λοιπόν ομοφωνία, όπως είπα, και θα ήθελα να επαναλάβω ότι οι αρμοδιότητές μας σε σχέση με αυτού του είδους τα θέματα είναι περιορισμένες. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν νομικές ρυθμίσεις οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους και διαφοροποιούνται ας πούμε και ε, στην Κροατία σαν παράδειγμα υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις διοικητικές για κατασχέσεις πολύ ψηλός αριθμός λόγω μη αποπληρωμής χρεών, ε, ε, λογαριασμών κτλ. Έχουν ε, λοιπόν ληφθεί αποφάσεις ε, εκατομμύρια φορές για τέτοιου είδους διαδικασίες, για την ενεργοποίησή τους. Ε, εκατομμύρια πραγματικά κάθε πολίτης ουσιαστικά εμπλέκεται. Το κόστος για τις διαδικασίες αυτές είναι πάρα πολύ υψηλό. Μιλάμε πολλές φορές για κατασχέσεις οι οποίες γίνονται ε, λόγω χρέους 300 ευρώ και η κατώτατη σύνταξη στην Κροατία είναι 300 ευρώ. Δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα λοιπόν λόγω ακριβώς των χρεών ε, τα οποία οδηγούν σε κατασχέσεις από πλευράς ε, αυτών που έχουν δανείσει, στους οποίους χρεωστούνται κάποια ποσά. στη Σλοβενία έχουμε διαδικασίες αντίστοιχες, ηλεκτρονικές όμως, κάτι το οποίο μειώνει το κόστος κάποιων δικαστικών διαδικασιών. Σε περιπτώσεις όπου η οικονομία δεν λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως η Κροατία, οι διαδικασίες που επιλέγονται λειτουργούν εις βάρος των πολιτών Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Κροατία, των οποίων οι λογαριασμοί έχουν μπλοκαριστεί. Εκατομμύρια εκατομμυρίων επαναλαμβάνω. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις επιτέλους οι οποίες θα επιτρέψουν την απλοποίηση των, της ζωής των πολιτών που έχουν ε, εις βάρος τους τέτοιου είδους διαδικασίες κατάσχεσης ε, προστατεύοντας φυσικά και τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Θα πρέπει οι διαδικασίες που θα επιλεγούν να είναι ταχύτατες, να επιτρέπουν την ανάκτηση των χρεωστούμενων ποσών τον ταχύτερο, με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο και να μειωθεί και το κόστος των διαδικασιών αυτών. όταν κάποιος κοστάει 300 ευρώ και οδηγείται σε ε, κατάσχεση, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάσχεση ακινήτου ε, και η διαδικασία αυτή κρατάει χρόνια ολόκληρα και στο τέλος το χρέος γιγαντώνεται και με τους μισθούς οι οποίοι υπάρχουν σε μια χώρα σαν την Κροατία δεν υπάρχει καμία λύση. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε κάποιες διαδικασίες ταχύτερες και αποτελεσματικότερες. Θα κάνετε κάποια πρόταση για αυτό το θέμα. Κύριε Μπούντα, για αυτό το θέμα ε, θέλετε ή για κάτι άλλο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να προσθέσω και άλλη ερώτηση. Μάλλον να ζητήσω από τον Υπουργό να μου απαντήσει την προηγούμενη ερώτηση για την προσχώρηση της Ρουμανίας στο Σέγγεν. Δεν μου απαντήσατε. Μία ερώτηση έκανα για το κράτος δικαίου και η δεύτερη ήταν για το Σέγγεν και την ένταξη της Ρουμανίας στο χώρο Σέγγεν. Δεν μου απάντησε ο υπουργό. Σας ευχαριστώ για την ε, ερώτησή σας. Ε, για το θέμα των εκτελέσεων κάποιων αποφάσεων αναφερθήκατε σε πολλά νομικά ζητήματα και στις συζητήσεις που γίνονται στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Κροατίας. Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Είναι περίπλοκο το θέμα, αλλά είναι εσωτερικό της Κροατίας. Έχει να κάνει με την κροατική νομοθεσία και βρήκαμε κάποιες λύσεις μέσα σε ένα πλαίσιο. Ορισμένες τις αναφέρατε εσείς, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την κροατική προεδρία ή μια διαδικασία ενιαία που θα μπορούσε να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη, ε, σε 28 κράτη-μέλη. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας είπαμε ότι ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προς όφελος όλων των πολιτών στην Ευρώπη. Για τα θέματα που τους απασχολούν εντός των αρμοδιοτήτων μας θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν κάποια συστήματα που είναι καλύτερα από κάποια άλλα και ορισμένα όχι και τόσο ιδανικά. Μπορεί να υπάρξει κάποια εναρμόνιση στο σύστημα επιβολής κάποιων αποφάσεων. Αλλά αυτό που ρωτήσατε είναι ενδοκροατικό ζήτημα. Προσπαθούμε να βρούμε καλύτερες λύσεις με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία για να λύνουμε καλύτερα τα προβλήματα. Πάντως δεν θα αφιστούμε προσπαθειών για να εργαστούμε προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών εγέννη. Για το ζήτημα του Σέγγεν και την ε, ερώτηση από τη Ρουμανία. Κύριε Μπούντα, θα πρέπει να ελέγξουμε πρώτα κατά πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ένταξη της ε, Ρουμανίας και η Κροατία αυτό το καιρό προσπαθεί να ανταποκριθεί στα προαπαιτούμενα και τα κριτήρια για να ε, ενταχθεί και εκείνη στον χώρο Σέγγεν. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ. Ε, καλή τύχη για το επόμενο εξάμηνο, πεντάμινο πια. Το 2007 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων διαπίστωσε ότι μόλις το 25% είναι τα μέλη στα διοικητικά συμβούλια ε, εταιριών γυναίκες. Ε, μεγάλων εταιριών. Αν δεν κάνετε τίποτα για τη στατιστική αυτή, δεν νομίζω να αλλάξουν και πάρα πολλά πράγματα τα ερχόμενα έτη. Είμαι ε, βέβαια ότι γνωρίζετε την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 ήδη και δεν θα σας πλήξει η ερώτησή μου. Προτίθεται η ε, Κροατική Προεδρία να λύσει αυτό το θέμα στο Συμβούλιο που είναι σε εμπλοκή για τη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εταιριών. Τι θα κάνετε για να κινητοποιήσετε, να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη, να ξεμπλοκάρουν το φάκελο. Και λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Ποια είναι η θέση της Κροατίας ε, γενικά για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Ποια είναι η θέση της χώρας σας και της κυβέρνησής σας, όχι της Προεδρίας και ποια ήταν το 2012. Υπάρχει λόγος που το ρωτάω αυτό. Γιατί είμαι από τις κάτω χώρες και το 2012 η χώρα μου και 13 ήταν αντίθετη με την πρόταση, ενώ τώρα το 2020 έχω λόγους να πιστεύω ότι είναι υπέρ και έχουν αλλάξει τα πράγματα στα κράτη-μέλη και θα βρείτε πλειοψηφία υπέρ της πρότασης. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποια είναι η θέση κρατικής κυβέρνησης, αν έχει αλλάξει τίποτα από το 2013 την παλιά θέση την ήξερα και την ξέρω, αλλά έχει αλλάξει τίποτα. Επίσης, τι θα κάνει η Προεδρία προς την κατεύθυνση αυτή για να κινηθεί το θέμα. Είστε αποφασισμένοι μετά από μια επταετία αδράνειας να προωθήσετε λίγο αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Όπως το είπατε άλλωστε, το 2017 υπό και Προεδρία έγιναν οι τελευταίες συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο για τούτη την οδηγία αλλά δεν υπήρχε ειδική πλειοψηφία για την έγκριση αυτού του κειμένου. Επομένως, ε, είναι μπλοκαρισμένο το ε, θέμα αυτό και δεν έχουν γίνει περαιτέρω συζητήσεις τα τρία τελευταία χρόνια. Το κείμενο είναι έτοιμο, αλλά για την ώρα ε, δεν έχουμε σημάδια που να δείχνουν ότι το θέμα αυτό θα προχωρήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Εμείς ως Προεδρία βεβαίως παρακολουθούμε την κατάσταση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και εάν ε, η ε, μειοψηφία ε, αλλάξει γνώμη, τότε ενδεχομένως θα ξανανοίξει το θέμα. Το πρόβλημα προέκυψε από την νομική βάση που είχε χρησιμοποιηθεί. Just a very short... Αν κατάλαβα καλά, γιατί ε, δεν είμαι σίγουρη. Εσείς θα κάνετε μόνο κάτι για το θέμα αυτό εάν και εφόσον ανοιχνεύσετε ότι η αναστέλουσα μειοψηφία δεν ε, υπάρχει πλέον, έχει αλλάξει γνώμη δηλαδή. Ε, και η Κροατία όπως και το 13 θα είναι εναντίον. Λοιπόν, λόγω της νομικής βάσης εμείς δεν υποστηρίζουμε την πρόταση και στα πλαίσια της Προεδρίας, λέω, παρακολουθούμε την κατάσταση. Αν εξελιχθούν τα πράγματα, θα παρέμβουμε. Ο Τίμο Βέλκεν. I'm listening. Ακούω, ακούω. Ακούω και προσέχω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα Έμεσα ε, θίξατε το θέμα του κράτους δικαίου, που είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της δικής σας Προεδρίας και δυστυχώς και των επομένων Προεδριών. Δύο ερωτήσεις έχω για το πρόγραμμα της δικαιοσύνης. Δύο από τους στόχους της περίοδο αυτής 2021-2027 είναι η διευκόλυνση και υποστήριξη δικαστικής συνεργασίας σε θέματα αστικά και ποινικά και η πρόθεση του κράτους δικαίου και δεύτερον να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η εκπαίδευση των δικαστικών έτσι ώστε να έχουμε ένα κοινό νομικό πολιτισμό και πολιτισμό κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Υπό την αίρεση βέβαια του PDP όλα αυτά. Τι ρόλο προτίθεστε εσείς να διαδραματίσετε στην εκπλήρωση αυτών των στόχων, πιο συγκεκριμένα. Τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε πολλές ανησυχητικές εξελίξεις σε διάφορα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία των δικαστικών συστημάτων. Μάλλον επιδεινώθηκε η κατάσταση. Ε, τι θα κάνετε ε, για να αποτρέψετε τέτοιες εξελίξεις στο μέλλον. Ιδιαίτερα τη στιγμή που ξέρουμε ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να τονωθεί ανάμεσα στα διάφορα δικαστικά συστήματα, ότι είναι αποτελεσματική δικαιοσύνη και αμερόληπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, στο πρόγραμμά μας αναφέραμε το γεγονός ότι το κράτος δικαίου ε, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Ε, γιατί άλλωστε μία από τις τέσσερις μεγάλες αρχές είναι το κράτος δικαίου και ε, η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Συνεργασία άνευ αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των συστημάτων, των υφισταμένων συστημάτων, ε, αυτών δηλαδή που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, αυτό θα ήταν κενό γράμμα. Επομένως, εμείς θεωρούμε απόλυτη προτεραιότητα το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα τον κανονισμό για το ε, αστικό δίκαιο, ε, είπα και προηγουμένως ότι το θέμα της ηλεκτρονικής κατάθεσης και αναγνώρισης των αποδεικτικών στοιχείων ε, είναι μεγάλης σημασίας γιατί με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί και η ε, προσβασιμότητα όλων των πολιτών στις διαδικασίες. Αλλά όσο δεν υπάρχει συμφωνία σε, στο υψηλότερο ε, επίπεδο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όταν στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο προκύψει συμφωνία, τότε και εμείς πολύ γρήγορα θα αναλάβουμε δράση ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Νομίζω πάντως ότι έχω ήδη απαντήσει ε, σε ερωτήματα σχετικά με το κράτος δικαίου και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για ένα από τα στοιχεία επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα από, μία από τις τρεις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Κυρία Μέλχιορ, uh, Χαίρομαι που είσαστε μαζί μας σήμερα, είναι μεγάλη χαρά. Και επίσης ε, είναι μια ευτυχή στιγμή αλλά και μια στιγμή δυσκολίας η ανάληψη μιας προεδρίας. Έχετε ένα τετραπλό σλόγγαν και ε, περιλαμβάνει τον όρο «Η Ευρώπη η οποία συνδέει». Ορισμένοι από τους συναδέλφους αναφέρθηκαν στο ότι υπάρχουν νομοθετικοί φάκελοι οι οποίοι έχουν κολλήσει πια στο Συμβούλιο για αρκετά χρόνια. Επιτροπολογία, γυναίκες σε υψηλές θέσεις, συλλογικές αποζημιώσεις. Εκτός αν μου διέφυγε κάτι, δεν αναφερθήκατε σε κάποια από τα σημεία αυτά τα οποία εκρεμούν στο Συμβούλιο. Δεν είναι προτεραιότητά σας. Θεωρείτε ότι είναι ανέφικτο να ξεμπλοκάρουν οι υποθέσεις αυτές. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, χαίρομαι που αναφερθήκατε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ελπίζω και οι συναδελφοί σας όλοι να προσυπογράψουν, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν το έχουν κάνει. Σχετικά με την ψηφιακή συνδεσιμότητα αναφερθήκατε και στο θέμα ε, των αποδείξεων ε, μέσω των δικτύων. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες οι οποίες είναι κάτι το οποίο μας αφορά ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αν θέλουμε μια ψηφιακά συνδεδεμένη Ευρώπη, μία από τις βάσεις είναι η ε, ασφαλής ψηφιοποίηση των δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αποδείξεις. Ε, ε, υπάρχουν τα θέματα λοιπόν των μεθόδων κρυπτογράφησης, της ασφάλειας της κρυπτογράφησης. Είναι θέματα τα οποία θα εξετάσετε. Έτσι ώστε να έχουμε λειτουργική κρυπτογράφηση άμεσα διαθέσιμη και για τις δημόσιες υπηρεσίες. Ένα από τα θέματα τα οποία επίσης ενδιαφέρει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μία πράξη ψηφιακών υπηρεσιών. Στα πλαίσια της πράξης αυτής προτείνεται να υπάρξει διάλογος γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και εμάς, αφορά τους πληθυσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πλατφόρμες, ε, η χρήση τους αυξάνεται όλο και περισσότερο και γι' αυτό θα πρέπει το σύστημα της δικαιοσύνης και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και των δικαιωμάτων των πολιτών να ε, μην μειωθεί μέσα από αυτές τις πλατφόρμες τις ηλεκτρονικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να πάρει μέρος στις, ε, στις ε, ακροάσεις με την Ουγγαρία για το κράτος δικαίου. Το Συμβούλιο το έχει αρνηθεί αυτό. Λόγω της σημασίας που έχει το κράτος δικαίου για την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς ως ε, ηγέτες σε αυτή τη φάση του Συμβουλίου, τι σημασία δίνετε στις ευρωπαϊκές αξίες. Θα φροντίσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριληφθεί και για το θέμα της Ουγγαρίας αλλά και για το θέμα της Πολωνίας όταν τεθεί. Έχετε θέσει πολλές ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη αν τυχόν δεν απαντήσω σε κάποια από αυτές. Τώρα για τα θέματα τα οποία έχουν μπλοκαριστεί όπως είπατε στο Συμβούλιο. Επιτροπολογία, συλλογικές αποζημιώσεις και προσφυγές, η θέση των γυναικών σε υψηλές διοικητικές θέσεις. Νομίζω ότι έχω δώσει κάποιες απαντήσεις ήδη μέχρι τώρα. Όπως είπα υπάρχουν προβλήματα διαδικαστικά σε κάποια θέματα. Σε κάποια άλλα θέματα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής βάσης. Ως εκ τούτου η Κροατική Προεδρία δεν έχει πολλές πιθανότητες να κάνει κάτι. Τώρα, για την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών. Εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τα θέματα της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και με τη μέθοδο των συλλογικών προσφυγών. Πρόκειται για κάποια σημαντικά βήματα προόδου, θα έλεγα, για τους καταναλωτές. Στόχος μας είναι να υπάρξει μια συμφωνία και με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της κρατικής προεδρίας. Η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου ήδη έχει γίνει και Ελπίζουμε να καταλήξουμε στους επόμενους μήνες σε μια συμφωνία για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Έχω, την όψη μου, έχω ε, τη χαρά να πω ότι η χώρα μου έχει επικυρώσει τη σύμβαση αυτή. Ως χώρα μέλος λοιπόν και ως χώρα που προεδρεύει στο Συμβούλιο θα συνεχίσουμε τον αγώνα εναντίον της οικιακής βίας, εναντίον της βίας εις βάρος των γυναικών. Και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και να καθοδηγήσουμε τις χώρες που δεν έχουν επικυρώσει. 21 χώρες έχουν επικυρώσει. Θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε και τις υπόλοιπες χώρες να το κάνουν, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον και το όφελος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης έτσι ώστε να προστατεύονται καλύτερα οι γυναίκες. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν εμπόδια στο συγκεκριμένο τομέα. Θα προχωρήσουμε στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για να επιτρέψουμε την επικύρωση της ε, Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από όλα τα κράτη-μέλη. Ε, τώρα για ο κανονισμός είναι σαφής. Ζούμε σε έναν κόσμο ψηφιακό. Τα πράγματα εξελίσσονται με υψηλότατες ταχύτητες. Υπάρχουν ε, λοιπόν κάποια ε, ε, θέματα ψηφιακά τα οποία δημιουργούν ορισμένες ερωτήσεις και πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες απαντήσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση. Αυτό ισούται με εξυγχρονισμό είναι βασική θα έλεγα πορεία προς την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την φάση προσπαθεί να καθορίσει το πλαίσιο, το διακανονιστικό και για το θέμα των αποδείξεων ε, σε επίπεδο ε, ψηφιακών συναλλαγών. Τώρα, για την κρυπτογράφηση και την ψηφιοποίηση ε, μεθόδων καταγραφής σε υπολογιστές κτλ. Και γενικότερα τη σχέση που μπορεί να έχει αυτό με θέματα που άπτονται του κράτους δικαίου. Ε, αναφερθήκατε στο θέμα της συμμετοχής του Κοινοβουλίου για την ακρόαση στο Συμβούλιο με την Ουγγαρία ή για την Ουγγαρία. Ήδη έχουμε πει ότι το Κοινοβούλιο είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο και θα συνεχίσουμε να αναφερόμεθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γύρω από τα θέματα ε, της Ουγγαρίας στις συζητήσεις του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον Υπουργό στην Επιτροπή μας και να σας ρωτήσω για το εταιρικό δίκαιο. Ελπίζω να είναι στη δική σας αρμοδιότητα, γιατί στη δική μας είναι. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη της Προεδρίας πολύ σύντομα θα καταθέσει ε, διάφορες προτάσεις για τη δέουσα επιμέλεια ε, στις επιχειρήσεις. Είναι προφανές ότι όλο και περισσότερο οι επιχειρηματίες ζητούν Ίσως κανόνες παιχνιδιού. Είναι πάρα πολλές εταιρείες που θέλουν να είναι υπεύθυνε να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, να είναι τμήμα της λύσης για το κλίμα, αλλά έχουν τον αθέμητο ανταγωνισμό ανεύθυνων επιχειρήσεων και διαφόρων ε, νομοθεσιών ε, όλο και περισσότερο ε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια διάφορες νομοθεσίες στις διάφορες χώρες και είναι μια ζούγκλα, δεν μπορεί κανείς να βρει το δρόμο του. Εσείς θα υποστηρίξετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτές τις προτάσεις και μάλιστα και προς νομοθετικές προτάσεις. Και δεύτερη ερώτηση που συνδέεται με την προηγούμενη. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την αναθεώρηση Ε, της ε, οδηγίας για την αναφορά ε, των εταιριών που επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια σε αυτούς τους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προχωρήσει και επίσης γνωρίζω ότι περιμένει και η Γερμανική Προεδρία να πάρει τη σκητάλη. Ε, γιατί το έχει αρχίσει η Φιλανδική Προεδρία. Η Κροατία όμως ε, και γεωγραφικά ακόμα είναι ένα πολύ ωραίο κράτος ανάμεσα στη Φιλανδία και τη Γερμανία. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά ε, τις επιχειρήσεις και το εταιρικό δίκαιο, βεβαίως θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Φυσικά είναι σημαντικό να δούμε και το θέμα της ε, ε, διακυβέρνησης όσον αφορά ε, τα θέματα αυτά. Ε, γιατί το ίδιο άλλωστε θα πρέπει να γίνει και για την αηφόρο ε, ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Ε, δηλαδή, οι επιχειρήσεις θα πρέπει στη διακυβέρνησή τους οπωσδήποτε να λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη αυτά τα θέματα. Άλλωστε υπάρχει και μία μελέτη η οποία αφορά ακριβώς το θέμα αυτό της διακυβέρνησης των επιχειρήσεων. Θα περιμένουμε λοιπόν την, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που θα πρέπει να προωθηθούν. βεβαίω, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωση στους τομείς αυτούς, αλλά νομίζω ότι ε, ο σωστό τρόπος είναι πρώτα να αποτυπούμε σωστά ε, τα στοιχεία και μετά να παίρνουμε μέτρα. Όσον ε, αφορά τώρα τις οικονομικές αναφορές, αναφέρθηκα στο θέμα αυτό και απαντώντας και σε μια άλλη ερώτηση Προς υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που εμποδίζουν τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων. Κυρίως ε, το πρόβλημα της νομικής βάσης ε, που δεν επιτρέπει την δημοσίευση αυτών των εκθέσεων η οδηγία για τις ε, συστάσεις ε, αναχώρα που είναι μοιρασμένη. Για τις επιχειρήσεις ε, στο country by country report είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τη δική μας και την Οικονομική Επιτροπή. Νομίζω ότι και οι υπηρεσίες της Κομισιόν θα ξέρουν τώρα πια πώς ε, μπορούν να σπρώξουν λίγο το θέμα έτσι ώστε να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις σοβαρά υπόψη της, τα non-financial reports. Αυτό, αυτή η νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική και ήδη υπάρχουν κάποια στοιχεία. το είναι ναι, ναι, πρόκειται για ένα ε, πολύ σημαντικό νομοθετικό κείμενο, αλλά επαναλαμβάνω θα πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση μαζί με όλους τους ε, εμπλεκόμενους και να δούμε. Η διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, ναι, είναι κάτι που μας απασχολεί και που οπωσδήποτε βρίσκει στο επίκεντρο των εργασιών μας ε, και μάλιστα θα διοργανωθεί και στην Κροατία μια διάσκεψη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Ομπρή. Euh, Καλημέρα κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Επιτρέψτε μου να επιμείνω στην ερώτηση που έθεσε ε, ε, η συνάδελφος όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια την οποία θα πρέπει να ε, επιδείξουν οι μεγάλες εταιρείες. Νομίζω ότι όταν μπερδεύεται τα έγγραφα, όταν μιλάμε για reporting non-financial και τα reports αναχώρα, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι λίγο ανησυχητικό, για να μην πω πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι τα μπερδεύεται. Θα σας τα πω από την πλευρά της Γαλλίας. Υπάρχουν κυβερνητικές οργανώσεις ε, στην Γαλλία που ελέγχουν ενώπιον της δικαιοσύνης την ε, Total ε, καθότι την κατηγορούν ότι είναι η εταιρεία η οποία εκλείει τα περισσότερα, το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα με τέτοιες εκπομπές δηλαδή σε ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως στην Γαλλία η οποία υπήρξε σκαπανέα αυτών των θεμάτων υπάρχει υποχρέωση δέωσης επιμέλεια ε, και εδώ δεν υπάρχει ακόμα, ενώ, όπως είπε και η κυρία Χαουτάλα προηγουμένως, ξεκινάει μια διαδικασία και ξεκινούν κάποιες διαδικασίες τέλο πάντων παρόμοιες σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα πρέπει να εκφραστείτε όσον αφορά το θέμα αυτό και όσον αφορά και την ευθύνη των ε, πολυεθνικών ε, ε, επιχειρήσεων. Σας επαναλαμβάνω ότι και εμείς περιμένουμε, αλλά και οι πολίτες περιμένουν, γιατί 100 μη κυβερνητικούς οργανώσεις έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, που είναι πραγματικά υποδειγματική και επομένως μπορείτε να βασιστείτε σε αυτά που έχει κάνει η Γαλλία για να προωθήσετε το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι που έχει ξεκινήσει αυτή η εργασία, αλλά αυτό που λέτε αδρανούμε μέχρι σότου κλπ. κλπ ε, δεν είναι δυνατόν ε, γιατί ε, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να καταρρεύσουν κτίρια όπως ας πούμε στο Μπαγκλαντές ή δεν ξέρω ποια άλλη καταστροφή να γίνει λόγω της αμέλειας που επιδεικνύουν οι διάφορε επιχειρήσει. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε σταυρωμένα τα χέρια. Τι θα κάνει η, Ευρωπα... η Κροατική Προεδρία έτσι ώστε να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο γίνεται πιο γρήγορα, τουλάχιστον να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα ε, τη μελέτη αυτή. Επίση, η Φιλανδική Προεδρία δεν είναι το αδρανή. Ε, έχει αφήσει έναν οδικό χάρτη όσον αφορά τα θέματα αυτά, άρα μπορείτε να ακολουθήσετε την οδό τη Φιλανδία. Θα το κάνετε και επίση θα διευκολύνετε ε, μια κοινή βάση συζήτησης με το Κοινοβούλιο μέσα. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι γι' αυτό. Ή, εν πάση περιπτώσει, το Συμβούλιο. je Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει συζητήσεις. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μέτρα σύμφωνα με συγκεκριμένα στοιχεία που θα έχουν προκύψει. Η Κροατική Προεδρία είναι απολύτως έτοιμη, είναι πανέτοιμη να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και να κάνει ό,τι χρειάζεται. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες που θα πρέπει και θέματα που πρέπει να σεβαστούμε. Κύριε τελευταία ερώτηση. Κύριε Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ως εισηγητής του σχεδίου οδηγίας για τις συλλογικέ αγωγές, ε, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι να προστατεύονται καλύτερα οι καταναλωτές απέναντι σε κάποιες ε, παρανομίες και εκτροπές των πολυεθνικών. Όλοι θυμόμαστε το Dieselgate ή την ακύρωση κάποιων πτήσεων Ryanair χωρίς καμία δικαιολόγηση. Όπως γνωρίζετε, στις 26 Απριλίου είχαμε ένα σχέδιο οδηγίας στο τέλος της περασμένης κοινοβουλευτικής περίοδου και το ψηφίσαμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. 579 ε, βουλευτές υπερψήφισαν. Έκτοτε ε, ξεκίνησε ο τριμερής διάλογος ε, στις 14 πρώτου στο Στρασβούργο. Συγχαίρω την Κροατική Προεδρία και σας το λέγω και το επιτελείο σας για το πνεύμα που πριτανεύει σε αυτές τις συνεδριάσεις. Ήμασταν πολύ επικοδομητικοί στις συνεδριάσεις. Αλλά μια που σας έχω εδώ, θα ήθελα να δω εσείς πώς το βλέπετε αυτό προσωπικά. Η Προεδρία διαρκεί ένα εξάμεινο. Ε, στο εξάμεινο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά περνάει και πολύ γρήγορα. Ε, σε ποιο βαθμό εσείς θεωρείτε ότι το κείμενο αυτό είναι απόλυτη προτεραιότητα για την Κροατική Προεδρία και αν θεωρείτε λογικό, ε, εφικτό και επιθυμητό να ε, καταλήξετε σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ. Ε, φυσικά, ο στόχος μας είναι να συμφωνήσουμε με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και φυσικά από πλευρά μα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε και το συγκεκριμένο φάκελο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, που ήρθατε να μας παρουσιάσατε τις ε, προτεραιότητες ε, της κρατικής προεδρίας. Είδατε πλήθος ερωτήσεων των συναδέλφων. Ορισμένες ερωτήσεις ήταν για συναφή θέματα και άλλες ε, ε, όχι, γιατί έχουν και τις προτιμήσεις τους και τα αγαπημένα τους θέματα τα μέλη της Επιτροπής μας. Και φυσικά αγωνιούμε να ξεπεραστεί η εμπλοκή στο Συμβούλιο. Και θα εκτιμούσαμε τα μάλλα οποιαδήποτε βοήθεια θα μπορούσατε εσείς να μας παρέχετε. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Έτσι με τόσο ακριβή τρόπο και εύστοχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις σας. Ζητώ συγγνώμη εάν δεν σας, ανικανοποίησα, δεν σας ικανοποίησαν όλες με απαντήσεις. Ε, θα φροντίσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Very much.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, στην ημερήσια διάταξη. Για την προσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών αγωγών. Λίγη ησυχία αν θα μπορούσαμε να έχουμε. Ένα θέμα μας έχει απομείνει. <laughs> Thank you. I would like to carry on with the meeting. So item 12 on our agenda. Θα ήθελα να συνεχίσουμε. Το ε, ε, μια 12 είναι για τις προσωπευτικές δράσεις για την προστασία ε, των ε, συλλογικών προσφυγών. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έγινε στις 14 Ιανουαρίου ενιστού είπαμε στην αρχή και ήταν η αρχή της διαδικασίας, θα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντιδιέ τον εισηγητή, για να μας πει τι διεμήφθηκε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και έχετε και το λόγο. Merci, Madame la et merci de Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για το κύρος που επιδείξατε και την πυγμή για να επικρατήσει εδώ ε, ησυχία. Πολύ ε, επιγραμματικά μας τα είπε ο Υπουργός, ε, μάλλον έτσι με υπεκφυγές απάντηση στην ερώτησή μου. Όπως σας είπα, στις 26 Απριλίου του 2019, την περασμένη θητεία εγκρίναμε κείμενο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 579 ψήφους και μάλιστα όλες οι πολιτικές ομάδες μαζί. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ε, υπερ και διακομματική. Αρχίσαμε λοιπόν τον τριμερή μας διάλογο στις 14 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο παρουσία του Didier Renders, του Επιτρόπου Δικαιοσύνης και της Κροατική Προεδρίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής ε, θέσαμε τρεις αρχές ως στόχους. Η πρώτη αρχή είναι η αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη των διαφόρων εισηγητών και τους ευχαριστώ για την ε, στράτευσή του γύρω από μια εντολή που είναι η εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω εδώ τη Λάρα τη Χάιντι, τη Μανό, ο Μπρί που δεν με ακούει αυτή τη στιγμή και τους υπολείπους και τον Ζήλ Λευγετό. Σας ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις συγητές και ξέρω ότι πέρα από τις διαφορές μας θα μπορέσουμε να βρούμε ένα δρόμο για να οικοδομήσουμε μια συνένεση. Εξάλλου αυτό είναι και το αντικείμενο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό έχουμε εκλεγεί και συνεδριάζουμε εδώ. Η δεύτερη αρχή είναι απαραίτητη αναζήτηση μιας σωστής ισορροπίας. Έχουν ε, θεμητές απαιτήσει οι καταναλωτές από τη μια και από την άλλη χρειάζονται και ασφάλεια δικαίου η επιχειρήσεις. Ανέκαθεν εγώ πίστευα ότι η οικονομία των επιχειρήσεων δεν είναι ο εχθρός της προστασίας των πολιτών. Και έχω καλέσει το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλους τους κοιόδης συγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να με παρακολουθήσουν σε αυτό το πνεύμα, που φυσικά απαιτεί από όλου κάποιες θυσίε. Η τρίτη αρχή είναι η επιθυμία να προχωρήσουμε γρήγορα. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ε, αρκετά φιλόδοξο έτσι, νευρικό, ε, δυναμικό, αλλά καθόλου εφικτό. Έτσι ώστε να καταλήξουμε μέχρι το τέλος της κρατικής προεδρίας. Βεβαίως, με την ησυχία μας θα τα δούμε τα θέματα, γιατί δεν έχει νόημα να βιαζόμαστε. Αλλά θέλουμε να εργαστούμε και γρήγορα. Έγινε ένας πρώτος τριμέρης διάλογος, πολιτικός. Ο δεύτερος θα γίνει στις 2 Μαρτίου. Μέχρι τότε θα έχετε φύγει δυστυχώς κυρία Πρόεδρε και όσους τριμερείς διαλόγους χρειαστούμε στο μεταξύ ανάμεσα στους δύο πολιτικούς. Λοιπόν, αλληλεγγύη γύρω από την εντολή μας, αναζήτηση δίκαιης και σωστής ισορροπίας και ε, βούληση ε, να προχωρήσουμε γρήγορα. Όλα αυτά τα συμφωνήσαμε στις 14 του μηνός. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι ανθόσπαρτα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, δυσκολίε, διαφορέ ανάμεσα στο κείμενο του Κοινοβουλίου και τη θέση του Συμβουλίου. Επίσης, υπάρχει και μια διαφορά που εκ πρώτης όψεως φαίνεται θεμελιώδης, αρκετά. Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να εναρμονίσει κάποια κριτήρια μόνο για τις διασυνοριακές υποθέσεις και όχι για τι εγχώριες. Το Κοινοβούλιο δεν το βλέπει έτσι, δεν το ψήφισε έτσι. Πάντως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα επαγρυπνούμε. Έτσι ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ως άλοθη, ως πρόφαση ε, ή ως ευκαιρία από το Συμβούλιο να ταλανίσει την ε, ευρωπαϊκή φιλοδοξία του κειμένου. Θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να ε, φτιάξει ένα σύστημα προσφυγών και να υπάρχει ένα συγκεκριμένος φορέας επιφορτισμένος με αυτό σε κάθε κράτος μέλος, ενεργός. Επίσης υπάρχουν διαφορές ως προς τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους αρμόδιους φορείς ε, για τις προσφυγές. Ποιος θα τους χρηματοδοτεί. Θα γίνει μια συζήτηση έτσι πολύ καθαρή και ειλικρινής ακριβώς για τη χρηματοδότηση και κάποιες αρχές χρηματοδότησης. Και δηλαδή εκείνος που θα χάσει ε, αυτή την αγωγή θα πρέπει να πληρώνει και τα δικαστικά έξοδα. Τα έξοδα της διαδικασίας. Αυτό με το οποίο διαφωνούμε με το Συμβούλιο είναι η προθεσμία μεταφοράς στην νομοθεσία. 42 μήνες έχει προτείνει το Συμβούλιο. Το θεωρώ τελείως υπερβολικό. Είναι σχεδόν τέσσερα χρόνια. Δηλαδή θα έχουμε ψηφίσει κάτι σε πρώτη ανάγνωση, στην περασμένη και όλα θητεία, για την αυξημένη προστασία των καταναλωτών, που θα τεθεί σε ισχύ μόνο στην επόμενη από τη θητεία. Εξ ονόματος του Κοινοβουλίου και των όσων εδώ ψηφίσαμε, το θεωρώ αυτό απαράδεκτο. Εμείς ψηφίσαμε μια λογική προθεσμία μεταφοράς και ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο, 12 μήνες είναι 6. Ένα μισό χρόνο αρκεί. Ε, δεν μπορεί να περιμένει η προστασία των καταναλωτών. Έχουμε πολλή δουλειά λοιπόν το επόμενο διάστημα. Θα αρχίσουμε την ενεργή τώρα διαπραγμάτευση. Εγώ θα είμαι ο εγγυητής ε, της εντολής που μου ανέθεσαν όλοι οι ευρωβουλευτές ε, πέρσι τον Απρίλιο με τόσο μεγάλη πλειοψηφία, αλλά θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε με ευφυΐα, με συνενετικό πνεύμα και ελπίζω. Κυρία Πρόεδρε, τώρα τα πρακτικά θα τα δείτε σε βίντεο, τι να κάνω. Ε, θα σας τα φέρω πάντως των επομένων τριμερών διαλόγων. Πάντως έχω βάσιμες ελπίδες και επειδή είμαι και φύση αισιόδοξο ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε μέχρι το τέλος της κρατικής προεδρίας. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αυτά τα οποία μας είπατε. Η κυρία Χάουταλα. Ε, Πράγματι εργαστήκαμε σε ένα καλό κλίμα. Ευχαριστώ τον κύριο Διντιέ για μια πραγματικά εξαιρετική προσπάθεια και πέτυχε ε, πολλά για το Κοινοβούλιο. Συνεχίσουμε να χαμογελάμε μετά την ολοκλήρωση του τριμερούς, του πρώτου τριμερούς διαλόγου και πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει σε κάποιο συμβιβασμό για το θέμα της ε, μεταφοράς ε, και της δημοσιοποίησης. Ε, όχι να περιμένουμε όμως το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου της τρέχουσας για να το πετύχουμε. Αυτό είναι υπερβολικό. Υπάρχουν ακόμα και το θέμα των διαφοροποιημένων οντοτήτων ομίλων, τα λεγόμενα split καταχωρισμένα ή, κατα... ή και χωρισμένα κριτήρια, και υπάρχει και το θέμα ότι οι μηχανισμοί αυτοί υπάρχουν σε ορισμένες χώρες και όχι σε όλες και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηριχθούν οι χώρες οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους μέσα. Υπήρξαν ιδέες μέχρι τώρα και διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά ήδη έχουμε σπείρει τους πρώτους σπόρους για ε, μια μελλοντική σοδιά ε, σε θέματα που δεν αφορούν αυστηρά τους καταναλωτές. Ε, πάντως είναι ένα πρώτο θετικό βήμα για την προστασία του καταναλωτή στην Ευρώπη. Χαίρομαι που ακούω θετικά στοιχεία για την προσπάθεια του συναδέλφου. Εγώ δεν πήρα μέρος στην προσπάθεια η οποία έγινε. Χαίρομαι για την συνεργασία η οποία διέκρινε όλους όσους πήραν μέρος. Επίσης ε, είναι σημαντικό να υπάρξει μια έκθεση πρωτοβουλίας και για τα hedge fund και για τις διαφορές και τις δυνατότητες διαιτησίας. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία ακόμα. Υπάρχει μια κάποια αισιοδοξία για το επίπεδο διαφάνειας το οποίο έχουμε ήδη πετύχει στο κείμενο στην φάση αυτή. Θέσατε ένα ερώτημα. Δεν κατάλαβα ότι ήταν ερώτημα, και ο κ. αλλά θα απαντήσω και στην ερώτηση που δεν κατάλαβα ότι ήταν ερώτηση. Υπάρχει πράγματα μια έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξαιρέσαμε το ότι οι συγκεκριμένες αυτές οντότητες μπορεί να είναι είτε δικηγορικές εταιρείες είτε και ταμεία, μία ε, χαρτοφυλάκια, όπως και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Είδαμε τι συμβαίνει στις Ηνωμένε Πολιτείες, είδαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αμερικάνικα συστήματα, είδαμε ακριβώς τα λάθη που έχουν γίνει και δεν θα τα επαναλάβουμε στην Ευρώπη και εγώ είμαι νομικός, είμαι δικηγόρος και ακριβώς εξαίρεσα τις δικηγορικές επιχειρήσεις από τη δυνατότητα να μπορούν ως δικηγορικές επιχειρήσεις να καταθέτουν α, συλλογικές αιτήσει αποζημίωσης. Μπορεί να το κάνουν εκ των υστέρων αυτό εφόσον οι πελάτες τους το κάνουν αλλά θα πρέπει μόνο συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών, αναγνωρισμένες ως τέτοιες, που θα μπορούν να καταθέτουν τέτοιες προσφυγές. Ομάδες για τις οποίες θα πρέπει να έχει υπάρξει ε, ε, διαφάνεια, θα πρέπει να έχει υπάρξει σωστή ενημέρωση για την ε, σύστασή τους, έτσι κανείς να μην μπορεί να στρεβλώσει και να προχωρήσει σε καταχρήσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, οι οποίες χρησιμοποιούν τις συλλογικέ προσφυγές για να αποσταθεροποιήσουν τις αντίπαλες εταιρείε τους, ενώ η πραγματική και μοναδικοί δικαιούχοι πρέπει να είναι οι καταναλωτές. Και ήδη είπαμε ότι όταν πάρα πολλοί α, ε, καταναλωτές μπορέσουν να ωφεληθούν από την αποκατάσταση της ζημίας τους, ακόμα και αν θεωρητικά αποζημιωθούν, ε, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα χρήματα, εφόσον υπάρξουν, θα δοθούν αποκλειστικά ε, προς όφελος ε, των καταναλωτών για τη δημιουργία σαν παράδειγμα ενός ταμείου αποζημίωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει από το α μέχρι το ω να μην υπάρξουν ε, ε, γεράκια είτε χρηματοπιστωτικά είτε δικηγορικά που θα εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που θα έχουν οι ε, προσφεύγοντες. Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. if I uh, um, something out of θα ήθελα να πω κάτι εκτός ε, ημερησίας διατάξεως. Ε. Ε, γιατί ούτω ή άλλω είναι έκτακτη η συνεδρία, να έχει και έκτακτο τέλο. Δεν ξέρω αν έχουμε τελειώσει, δεν ξέρω αν θέλετε πρώτα να τελειώσετε το τη και μετά να μου δώσετε το λόγο. Όπω θέλετε, παρακαλώ. Να ασκήσετε το δικαίωμα του Πρόεδρου. Έχουμε ένα τελευταίο θέμα. Ανακοίνωση των συντονιστών. Και θα ήταν κρίμα να μην το κάνουμε κι αυτό. Ήταν εξαιρετική η συνεδρίαση των συντονιστών σε φιλικό κλίμα. Αποφάσισα λοιπόν να αποσύρουν το αίτημα για η ε, ε, ε, έκθεση ίδιας προβουλίας όσον αφορά ε, την, ε, την ε, περίοδο 17-18 όσον αφορά την αμοιβαιότητα και την αναλογικότητα και να το κάνουν αργότερα. Να εξηγήσουμε ότι ο λόγος είναι ότι μας πρότεινε η ΦΑΜ μια κοινή έκθεση νομοθετικού περιεχομένου και επομένως έπρεπε κάτι να βγάλουμε από αυτό το τρίμηνο και να το προσθέσουμε αλλού. Αποφασίστηκε λοιπόν να, η κύριοι Ζαμπράσκη, ε, όσον αφορά τον κύριο Πουσδεμόνα και την ασυλία του και τον κύριο, την ασυλία του κύριου Κομίνα. Services Act adapting commercial and civil rules for the commercial entities operating online. Mr. Del... Del Blanco, για έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, για το, πλαίσιο, ε, για το ηθικό πλαίσιο ΙΑΙ, ο κύριος Βόσα. Ε, για το ε, θέμα της αστικής ευθύνης, ο κύριος Λεμπρετών επίσης για θέματα ερμηνείας διεθνών ε, κανόνων, ο κύριος Σέσνε για την ενδιάμεση έκθεση για την πνευματική πρωτοβουλία, Σαβρίνα Πίτσον τίλι, την New σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του ενωσιακού δικαίου. Το κρατάει, κρατάει την έκθεση αυτή. Ο κύριος Μπράγερ, εισηγητής ε, γνωμοδότησης ε, ΙΜΚΟ για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Επίσης, ε, ε, δώσαμε άδεια για την ενεργοποίηση του άρθρου, της διαδικασίας του άρθρου 78 ε, μαζί με την ΦΑΜΑ, καθώς επίσης και πρόγραμμα το, του, δικαστηρι... του ελεγκτικού συνεδρίου για το Non-Financial Reporting Δεν νομίζω ότι έχω να πω τίποτα άλλο σε σχέση με τους συντονιστές, επομένως ευχαριστώ πολύ και σας δίνω το λόγο. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ γιατί εγώ ανέλαβα την θλιβερή αυτή, ε, το θλιβερό αυτό καθήκον να σας αποχαιρετήσω σήμερα. Δεν είναι λυπηρό μόνο ε, γιατί υπάρχει ένα ειδικό πολιτικό πλαίσιο ε, στο οποίο όλα αυτά συμβαίνουν αλλά και γιατί μας άρεσε πάρα πολύ να δουλεύουμε μαζί σας είστε ευφυείς, ε, είστε πραγματικά εξαιρετικοί. Βλέπω ότι οι διάφοροι φεύγουν, υπάρχει κινητικότητα, εν πάση περιπτώσει είστε και ένα άτομο το οποίο ε, πραγματικά ε, μας οδήγησε σε ασφαλή ύδατα χωρίς, χωρίς, πολλές, χωρίς πολλές αναταράξεις. Πραγματικά σας εκτιμήσαμε ε, και είναι πάρα πολύ λυπηρό που ολοκληρώνεται έτσι αυτή η διαδικασία. Ε, η ομάδα μου θα ήθελε πραγματικά να συνεχίσει η παρουσία σας εδώ και νομίζω ότι λέγοντάς το αυτό εκφράζω και την άποψη των ε, άλλων συναδέλφων. Σας ευχαριστούμε για όλα και για να σας δείξουμε την εκτίμησή μας από εμά και από τη Γραμματεία ένα μπουκέτο με λουλούδια μπορείτε να πάρετε μαζί σας. Γιατί ελπίζω να ξαναέρθετε να μας δείτε και είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή δεν θα ξαναέρθετε μόνο για να μας επισκεφτείτε, αλλά θα ξαναέρθετε ως μέλη. Presidente, anche io voglio associarmi θα ήθελα και εγώ να, με τη σειρά μου να εκφράσω την συμπάθεια, τις ευχαριστίες και την εκτίμησή μου στο Πρόεδρο της Πρόεδρου. Ε, εμείς προερχόμαστε ο καθένας από διαφορετική πολιτική ομάδα. Αλλά ε, δημιουργούνται συμπάθειες, καλή συνεργασία ε, και έστω και αν έχει κανείς διαφορετικές πολιτικές απόψεις, είναι πάντα λυπηρό να μην έχει κανείς ε, να συνεργάζεται με μια τέτοια πρόεδρο. Θα ήθελα λοιπόν για μια φορά ακόμα να επαναλάβω την εκτίμηση που τρέφω στο πρόσωπό σας. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή στην πολιτική μας πορεία θα ξανασυναντηθούμε και πραγματικά σας εύχομαι τα καλύτερα για τη μελλοντική σας καριέρα. Um, I like to say thank you so Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά να ε, προεδρεύω σε αυτή την Επιτροπή. Το ευχαριστήθηκα, ευχαριστήθηκα κάθε στιγμή της Προεδρίας. <laughs> So it, it was, it's been quite challenging. Ε, κοιτάξτε, εμένα μου δώσανε το βραβείο του πιο καλού μαθητή, αυτού που μαθαίνει περισσότερο από όλους και με ταχύτητα. Ε, λυπάμαι όμως που δεν κατάφερα να μάθω καλά γαλλικά. Εντάξει, μπορώ να το... θα μπορούσα να είχα κάνει μια προσπάθεια να πω τουλάχιστον ευχαριστώ και γεια σας. Σας λέω λοιπόν au revoir στα γαλλικά και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Και σίγουρα θα παρακολουθώ τι γίνεται, τις εξελίξεις με τις ε, εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας. Θα, οπωσδήποτε θα μετρώει περιέργεια να μάθω τι γίνεται.